βοηθήσουν πολύ αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα ε, και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αλλαγή ε, προοπτικής των Ελβετών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα, αν με επιτρέπεις Δόρης, να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ θερμά όχι μόνο για τη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά για τον ενθουσιασμό σου, για τη δουλειά σου και να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση στη Μαδρίτη το Σαββατοκύριακο που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Lux. Στις 17 δεν θα είμαι δυστυχώς εκεί, αλλά 18 και 19 θα συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις εκδηλώσεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Και πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ανάγκη από κόσμο σαν την Doris Pack για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα στο έργο μας, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι και έχουμε ανάγκη. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει σε μια μισή ώρα περίπου. Θα ξεκινήσουν στι 12 οι ψηφοφορίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, που είναι και το τελευταίο. Διαφορετικό αυτό το θέμα βέβαια. Είναι μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευεξή την καλή μεταχείριση των οτόκων ορνήθων μία προφορική ερώτηση από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου. Συντάκτη τη προφορική ερώτηση είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία, ο κύριος Δεκάστρο, που έχει το λόγο για πέντε λεπτά για να υποβάλει την ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να εξετάσουμε ένα θέμα στρατηγικής σημασίας, το θέμα της ευεξίας των ζώων στην Γεωργία. Την 1η του 2012 θα τεθούν σε ισχύ τα κριτήρια της οδηγίας 74 ε, του 1999 για την ε, μεταχείριση των ατόκων ορνήθων και την απαγόρευση των μη διευθετημένων κλοβών. Οι μη διευθετημένες κλοβοί θα απαγορεύονται πια στην πτηνοτροφία. Έτσι θα εξασφαλίσουμε καλύτερη μεταχείριση των οτόκων ορνήθων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο Γεωργίας του Ιουλίου του 1999 ήταν ένα πολύ σημαντικό συμβούλιο και μια ημερομηνία ορόσημο γιατί τότε ο Υπουργό Γεωργίας συμμετείχα σε εκείνο το Συμβούλιο Υπουργών και υπερψήφισα αυτή την οδηγία. Ένα χρόνο μετά διαπιστώνουμε ότι οι γεωργοί, οι πτηνοτρόφοι αρχίζουν και προσαρμόζονται σε αυτές τις ε, υποχρεωτικές, ε, αλλά δυσεφάρμοση μερικές φορές ε, διατάξεις. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά μόνο την ευεξία των ζώων, αλλά και την ευημερία των γεωργών που προσπαθούν να εφαρμόσουν την οδηγία 74 του 1999. Και για να επιτύχουμε εναρμονισμένη εφαρμογή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου και την αποφυγή του ανταγωνισμού στην αγορά αυγών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και αυτό και το θέσαμε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Γεωργίας. Τους τελευταίους μήνες έγινε πολύ σημαντική συζήτηση και έντονο έργο με τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων που κατέληξε στην προφορική ερώτηση της 28ης Οκτωβρίου. Θέτουμε πολύ σημαντικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, τι μέτρα θα προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Τι δράση αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους όρους της οδηγίας. Τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των φτηνοτρόφων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία ή τι μέτρα θα πάρει η Επιτροπή για να παρεμποδίσει ενδεχόμενο αθέμητο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά αυγών, γιατί οι τρίτες χώρες δεν είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν την ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέσαμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε τις απαντήσεις της περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει διαφάνεια στην αγορά αυγών, αμοιβαιότητα των κανόνων και καλύτερη σύγκληση των διεθνών κανόνων σε ό,τι αφορά την ευεξία και την σωστή μεταχείριση των Είναι ένα θέμα που μα απασχόλησε στην Επιτροπή Γεωργία από την αρχή τη κοινοβουλευτική μα θητεία. Το θέμα αυτό είναι θεμελιώδη σημασία γιατί ζητούμε τεράστιε προσπάθειε και πολύ δύσκολε από του δικού μα γεωργού κτηνοτρόφου και πτηνοτρόφου, αλλά θα πρέπει και η αγορά να αναγνωρίζει αυτού του κανόνε και φυσικά να μην ε, ε, δημιουργούνται συνθήκες σε θέμα του ανταγωνισμού που θα φέρνουν σε δυσμενή μοίρα τους δικούς μας ντόπιου γεωργούς και κτηνοτρόφους. Θα πρέπει αντίθετα ο σεβασμός των κανόνων της οδηγίας να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα για τους δικούς μας παραγωγούς. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επίτροπος Βασιλείου για να απαντήσει στον κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Καταρχήν θα ήθελα να σας μεταφέρω τη συγγνώμη του Επιτρόπου Ντάλη που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί αυτό προσώπος, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον αντικαταστήσω εγώ απαντώντας στην προφορική αυτή ερώτηση για την ευεξία των ζώων. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η απαγόρευση των συμβατικών συστοιχιών κλωβών που υιοθετήθηκε το 1999 συνιστά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σημαντική βελτίωση ό,τι αφορά την ευεξία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εκ τούτου η απαγόρευση αυτή έδωσε λαβή για σφοδρέ ε, και συναρπαστικέ συζητήσει ε, παντού στον κόσμο. Τα κράτη-μέλη είναι ε, τα αρμόδια για την εφαρμογή τη νομοθεσία ότι αφορά την προστασία των οτόκων ορνήθων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να παρακολουθήσει την συμμόρφωση των κρατών μελών με την οδηγία αυτή και μάλιστα μερικέ φορέ διοργανώνει ελέγχου και επιθεωρήσεις ε, που διενεργούνται από τους ε, εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα στοιχεία που ετησίως χορηγούν τα κράτη-μέλη γίνεται αυτός ο έλεγχος σε συνδυασμό με τους ε, ελέγχους που γίνονται και στα αγροκτήματα. Πέρυσι, ε, μάλιστα τον περισμένο μήνα τα επίσημα στοιχεία ε, των κρατών μελών υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από 24 ε, χώρες μέλη ό,τι αφορά τις συνθήκες ε, που επικρατούν στους κτηνοτροφικούς σταθμούς. Μέχρι στιγμής όμως μόνο 18 κράτη-μέλη υπέβαλαν τα πλήρη στοιχεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 66% των χώρων παραγωγής σε αυτά τα 18 κράτη-μέλη εφαρμόζουν συστήματα ελευθέρας βοσκής για τις οτόκες όρνηθες. 29% ε, με ε, τα συστήματα της απαγόρευσης, 3,9% με συμβατικές κλοβούς και ε, ένα μικρό ποσοστό με άλλο είδος κλοβών. Πάντως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλά κενά στα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη και μάλιστα τρεις χώρες μέλη δεν έδωσαν κανένα στοιχείο, ενώ έξι χώρες έδωσαν μόνο μερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους παραγωγής. Οπότε η εικόνα που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πλήρης και μάλιστα εξακολουθούμε να ε, οχλούμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που μας χορηγούν και μάλιστα και στη μόνιμη επιτροπή της ε, αλυσίδας τροφίμων και υγείας των ζώων ε, κάνουμε τέτοιες εκκλήσεις καθώς και στην συνεδρίαση των αξιωματούχων κτηνιάτρων. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κατά πόσο εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην εξασφάλιση ε, των μέτρων που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη προκειμένου εμπρόθεσμα να απαγορεύσουν τις μη διαθετημένες κλωβούς. Και μάλιστα τα αυγά που δεν παράγονται ε, με βάση τις διατάξεις για την προστασία των οτόκων ορνήθων δεν είναι εμπορεύσιμα νομίμως με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Βέβαια, μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης ε, θα δημιουργηθεί του χρόνου μετά την συνάντηση των ενδιαφερομένων που θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2011. Τότε θα διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης. Σήμερα η εισαγωγή των κελίφων αυγών είναι πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό και εφαρμόζονται ε, τα, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, υγείας. Και μάλιστα οι συσκευασίε που περιλαμβάνουν αυγά εισαγόμενα από τρίτε χώρε, όπου δεν υπάρχουν σαφή εχέγγυα για την αντιστοιχία των ε, προδιαγραφών παραγωγής μετακινητικά, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σήμα ε, μέθοδοι πτυνοτροφίας ε, μη συμβατή με τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Με το σήμα αυτό θα γίνεται σαφή διάκριση μεταξύ των εισαγόμενων αυγών που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και των εισαγόμενων αυγών που τις πληρούν. Ε, Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους στη συνάντηση που, όπως σας είπα, θα λάβει χώρα στις 19 Ιανουαρίου του 2011 στις Βρυξέλλες και εκεί θα εξεταστούν διάφορες εναλλακτικέ μέθοδοι προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή ε, συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στους εκπροσώπους των ομάδων εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα λάβει Πρώτα το λόγο η κυρία Εστέρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τελικά ταχύτατα προχωρούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία τα προϊόντα για τα οποία συζητάμε δεν θα ε, ε, ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το 30% των αυγών ε, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι ευρωπαϊκά αυγά. 8 με 13% των αγροτών, των πτηνοτρόφων έχουν προβλήματα ε, για να αντιμετωπίσουν ε, την ε, παραγωγή αυτή σύν το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν πολύ ακριβά τα αυγά ελε, ελευθέρας βοσκής ε, είναι πολύ πιο φτηνά τα άλλα πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και μη λέτε τώρα ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται ε, και υπεύθυνα είναι τα κράτη-μέλη. Εμείς προσβλέπουμε σε εσάς ε, κυρία Επίτροπε ε, γιατί πραγματικά δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που αποφασίστηκαν. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση, ζητούμε να απαγορευτούν οι συστοιχίες ε, ζητούμε να δια να αλλάξουν κανόνες κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, προβλέπουν τέτοια απαγόρευση. Ε, εδώ πιστεύω ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Κομισιόν, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Ντελάνγκη. Για ένα λεπτό το λόγο έχει εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών, ο κύριος Καπόλας Άντος. Eh, Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και ο κύριος Δεκάστρο, ως Υπουργός Γεωργίας τότε, πριν από 12 χρόνια, συμμετείχα στην ε, συζήτηση και στην έγκριση της οδηγίας που εξετάζουμε εκεί. Θυμάμαι ότι ήταν μια χρονοβόρα συζήτηση και πολύ δύσκολη, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο συγκρόμενες αξίες. Να εξασφαλίσουμε την ευεξία των ζώων, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η λύση που βρήκαμε έδωσε έμφαση στην ευεξία των ζώων και στην χορήγηση μια αρκετά μακροχρόνια μεταβατικής περίοδου στον παραγωγό για να προσαρμοστεί. Παρόλο που έχει περάσει καιρό που εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες, ε, η έλλειψη ε, πλήρων στατιστικών στοιχείων μα δημιουργεί προβλήματα, όπως είπε και η κυρία Επίτροπος. Γιατί κάποιες επιχειρήσεις που επενδύουν και κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να συμμορφωθούν με την οδηγία θα πρέπει να πλήττονται και να γίνονται θύματα της, του αθέμητου ανταγωνισμού από άλλους παραγωγούς που δεν σέβονται αυτές τις προδιαγραφές. Θέλουμε πολύ πιο λεπτομεριακή ανάλυση για να δούμε πώς ακριβώς έχει κατάσταση στα κράτη-μέλη. Και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την οδηγία αυτή από την 1η Πρώτη 2012. Επίσης, πώς μπορούμε να μάθουμε αν υπάρχει ένα ε, ελάχιστο εναρμονισμένο πλαίσιο κυρώσεων μεταξύ των κρατών μελών που να επιβάλλεται στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Αυτά και θα ήθελα να σας εκφράσω για την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ε, θα ζητήσουμε τα σημεία F8, 9 και 14 θα τα καταψηφίσουμε γιατί οι στόχοι τους είναι αμφιλεγόμενοι σε ό,τι αφορά την συμβατότητα με την οδηγία και δεν νομίζω ότι θα συνάδουμε με την αξιοπιστία της ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος George Lyon εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Δύο λεπτά. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπε, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που δώσετε στην αρχή της συζήτηση. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι άσχετα από το κατά πόσον έχουμε πλήρη υποπτική εικόνα της κατάστασης το γεγονός είναι ότι από πρώτου του 2011 80 εκατομμύρια αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράγονται με παράνομο σύστημα δεν πρόκειται ε, να αλλάξουν τα πράγματα μέχρι τότε βεβαίω. Δεν πρόκειται να προλάβουμε να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή. Η παραγωγή ε, στην Ευρώπη, τουλάχιστον να μιλήσω για τους ε, παραγωγούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ξοδέψει δύο εκατομμύρια ο καθένας για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο καινούριο σύστημα. Τι να τους πω τι να τους πούμε, τι να τους πούμε, τι να πούμε επίσης τους καταναλωτές ότι που τους έχουμε πει ότι δεν θα παράγονται αυγά, δεν θα κυκλοφορούν στην αγορά αυγά τα οποία θα παράγονται στις συστοιχίες κλοβών. Τι, τι θα πούμε σε αυτούς τους οποίους είπαμε επανειλημμένως ότι ε, θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν οι κανόνες, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Ε, ε, ε, ε αυτοί που προσαρμόστηκαν θα πρέπει τα κράτη-μέλη των οποίων παραγωγή και καταναλωτές προσαρμόστηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να επιβραβευθούν θα πρέπει να μην γίνουν θύματα της κατάστασης θα καλύτερα θα ήταν να φτιάξουμε ένα κατάλογο και να δείξουμε με το δάχτυλο ακριβώς αυτούς που δεν προσαρμόστηκαν. Λοιπόν, θα πρέπει κυρία Πρόεδρε να μας δείξετε κι εσείς να πείτε κι εσείς και να δείξετε ένα σήμα να κάνετε ένα ε, σήμα σε όλους ότι κατανοείτε την κατάσταση και θα φροντίσετε να τη διορθώσετε Για 3,5 λεπτά το λόγο κύριος Μάρτιν Χάουσλινγκ εκ μέρους των Πρασίνων Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε δεν μας έπεσαν αυτά που είπε η Κομισιόν στο... Επιτροπή. Δεν ήταν ιδιαίτερα πιστικά. Το είπε ο κύριος ε, Σαζάη ότι το πρόβλημα θα το έχουμε το 2012 και το 2013 που τα αυγά θα φτάσουν να είναι παράνομα στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν επίκειται κάποια παραβίαση των συνθήκων. Θα πρέπει να ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους τους γεωργούς και τους ε, αυγοτρόφους και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη. των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προστασία των ε, ε, των ζώων και γι' αυτό θέλω να τονίσω γιατί εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θελήσαμε να έχουμε μια υψηλότερη προστασία σε σχέση με τις συνθήκες εκτροφής των ορνήθων. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τώρα τι θέλει να κάνει η Κομισιόν. Εμείς έχουμε ζητήσει ήδη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να γνωρίζουμε. Θα θέλαμε να ξέρουμε από την πλευρά τη Κομισιόν ποιε είναι οι προτάσει που θέλει να διατυπώσει. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να συζητείτε και το να παρατείνουμε τις προθεσμίες. Εγώ το θεωρώ απόλυτα απαράδεκτο να τιμωρούνται ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι έχουν εφαρμόσει τις αυστηρότερες προδιαγραφές και όλοι οι άλλοι να έχουν το δικαίωμα με μεταβατικές περιόδους να συνεχίσουν να εκτρέφουν όρνηθες και αυγά κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Αναφερθήκατε στο θέμα της σήμανσης. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα προϊόντα που περιέχουν αυγά και γίνονται από φρέσκα αυγά. Πώς μπορούμε να, να έχουμε σήμανση των προϊόντων από λεύκομα αυγού, παραδείγματος χάρη. Και είπαμε, μέχρι 10 χρόνια είναι ο χρόνος για την αποθήκευση των αυγών. Θα πρέπει να γνωρίσουμε όλοι ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή, αυτό το χρονικό διάστημα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητε εξαίρεση για οποιοδήποτε κράτος μέλος. Και δέκα χρόνια πράγματι επαρκούν. Έχουμε μια πρωτοπόρο θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τα θέματα προστασία των οτόκων ορνήθων. Εμείς έχουμε αυτό το επιχείρημα πάντα έναντι των πολιτών και καταναλωτών και φυσικά και το Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξουν την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Επομένω, να, θα πρέπει να αναλάβει δράση η Κομισιόν και δεν θα πρέπει να αφήσει να διαιωνίζεται μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου ικανοποιητική, δηλαδή να περιμένουμε το 2012. Ευχαριστώ πολύ από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ Έχει το λόγο ο κύριο James Nicholson για δύο λεπτά. Διότι ένας από τους ε, από τους συντρόφους του και συγκομματικούς του έχει απαρνηθεί το δικό του ένα λεπτό. Δύο λεπτά έχετε κύριε Νίκολσον. Πρώτα απ' όλα. Εγώ δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν σήμερα. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις όπου οι αρμόδιοι της Επιτροπής ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και αυτά που μας είπαν δεν ήταν μονάχα απαράδεκτα, ήταν αβυσαλέα χαμηλό το επίπεδο, ήταν ένα έσχος για να το πω έτσι. Εγώ άκουσα αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα, αλλά η Επιτροπή δεν μας έχει δώσει τίποτα περισσότερο από μόνο την πρόταση να γίνει μια συνάντηση των εμπλεκομένων τον Ιανουάριο. Τι θα πείτε λοιπόν στους εμπλεκόμενους, τι θέλετε, να επιτύχετε με μια τέτοια συνάντηση. Πρέπει να καταλάβετε σήμερα ότι και οι τελευταίες κότες οι οποίες βρίσκονται στις παραδοσιακές, στους παραδοσιακούς κλωβούς θα πρέπει να βγουν από εκεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε συμβατικούς κλωβούς. Ίσως μπορείτε να πείτε περισσότερο λέγοντας ότι τα αυγά από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν διαφορετική σήμανση. Μα τι εννοείται με αυτό θα αποδεχθείτε το γεγονός ότι τα αυγά που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο παράνομο, δηλαδή από μη επιτρεπόμενους κλοβούς, δεν θα επιτρέπεται να εξάγονται από τη χώρα παραγωγής τους και δεν θα μπορούν να την χάνουν εμπορίες. Έχουμε πρόβλημα. Όπως είπε ο Τζορτζ Λάιον, έχουμε 83 εκατομμύρια αυγά, τα οποία θα είναι παράνομα την 1η Ιανουαρίου 2012. Τι θα γίνει με ο κόσμος ζητάει να φάει αυγά με λάτα ή σφιχτά. Πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουμε προς τα που κινούμεθα. Θέλω να μας δώσετε μια διαβεβαίωση ότι θα έρθετε ενώπιον του Κοινοβουλίου το Μάρτιο και θα μας δώσετε σωστές προτάσεις σε σχέση με αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε για να εξασφαλίσετε μια κατάσταση η οποία θα είναι ελεγχόμενη και όχι μια κατάσταση που θα είναι ομελέτα. Διότι πάρα πολλοί έχουν πληρώσει εκατομμύρια για να τροποποιήσουν του κλοβού του. Δεν μπορούν τώρα να πληρώσουν την ύφη για του άλλου οι οποίοι δεν έχουν τήρηση στι προδιαγραφές. Ευχαριστώ Τζιμ για την Ευρώπη τη ελευθερία και τη Δημοκρατία, Για δύο λεπτά και μισό έχει ο κύριο Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γέννησε αυτήν την κρίση. 100 εκατομμύρια από αυτέ τι όρνηθε θα συνεχίσουν να βρίσκονται στου κλοβού και δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα επιμελητία. Το θέμα είναι το πώ θα εφαρμοστούν αυτέ οι διατάξει. Ε, τελικά, επειδή κατέχει τη θέση το Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισθάνεται περήφανο, όμω ε, έτσι θα έχει πληγεί πάρα πολύ ο κλάδο στην χώρα μα. Για να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε. Ε, σε 24 ώρε 100 εκατομμύρια ε, ε, κότες, τι πώς θα εξαφανιστεί και τι θα γίνει με, θα τα κάνει το ομελέτα 83 εκατομμύρια αυγά μέσα σε μια μέρα τι θα κάνει ο καταναλωτής, τι θα κάνει με αυτά τα 83 εκατομμύρια αυγά κάθε μέρα θα πάνε στην Ουκρανία, στην Ινδία, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή ε, και μέσα σε, σε αυτού του είδους ε, τις συστοιχίες των κλοβών θα έχουν δημιουργηθεί αυτά τα αυγά και αυτό θα έχει πάρα πολλές συμβολές για την υγεία πρόκειται λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος να διαδοθεί αυτή η πρακτική, δεν μπορεί να τη φρενάρει κανείς και θα έχουν ε, προβλήματα η παραγωγή στην χώρα μας και οπότε και τρόπο είναι σαν να ε, διώχνουμε τη βιομηχανία μας οπότε ε, θα χρειαστούν επίσης και πάρα πολλά έξοδα για την συμμόρφωση εγώ νομίζω ότι αυτό είναι θνησιγενές σαν ιδέα δεν είναι δυνατόν να να περάσει και επίσης θα υπάρξουν στάσεις στον ΠΟΕ άρα θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις σε κάποιους που θα πρέπει να αργήσουν να συμμορφωθούν αλλά δεν μας ε, αρέσει το ότι έχουμε αυτή την εικόνα των αυγών που το 2012 πρόκειται να μην έχουν τη σχετική ένδειξη και σφραγίδα ε, και αυτά θα εξάγονται εμείς πάντοτε είχαμε κάποιους κωδικούς που χρησιμοποιούσαμε και αυτό δήλωνε τον τρόπο παραγωγής κλπ. Αυτή η διαδικασία γίνεται εδώ και τώρα που μιλάμε και στη δική μου τη φάρμα και έγινε αξιόπιστη η μέθοδος. Η Κομισιόν το βρίσκει πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να οργανώσει κάτι αντίστοιχο ε, παρά το ότι αυτό χρειάζεται. Οπότε βεβαίω. Πρόκειται για την ίδια επιτροπή η οποία αναγκάζει τους ε, προβατοπαραγωγούς στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουν τη σχετική σήμανση πάνω στα αρνιά. Ε, Επομένω, το, το, το έλασον κακό είναι να δώσουν παρεκκλήσεις και να έχουν κάποια ε, περιθώρια κάποιες χώρες όσον αφορά αυτή τη σήμανση. Και επίσης θα γίνεται και κάποιο είδους επιθεώρηση και να υπάρχει μια βάση δεδομένων όσον αφορά αυτούς που έχουν τις συστοιχίες των κλοβών γιατί οι περισσότεροι στο λιανεμπόριο ε, συμμορφώνονται όσον αφορά την ημερομηνία λήξη, αλλά για να τηρηθεί η ξύλινη πρέπει να υπάρχει σήμανση αντίστοιχη στα αυγά. Ευχαριστούμε, συνάδελφε πρόεδρος Και τώρα τελειώνει αυτή η φάση του, του συζήτηση και το λόγο θα τον λάβει για ένα λεπτό ο κύριος ε, Ματράς από τους μη εγγεγραμμένους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για κάτι που δεν αφορά μόνο τις ε, κότες και τα κλουβιά, αλλά είναι το θέμα το κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να, να τι θα σέψει την, την αγορά, γιατί ε, μέχρι το 2012 θα έχουν θα έχουμε φτάσει σε κατάσταση παρανομίας για όλα τα προϊόντα ε, γιατί κάποιοι οι χώρες του Βορρά έχουν ε, συμμορφωθεί, όλοι μας έχουν και μεγάλο παραγούς οι οποίοι αρνούνται να συμμορφωθούν, αυτό σημαίνει τεράστιες δαπάνες ε, και επίσης δάνεια. Έχουμε, εδώ λέει εδώ πέρα ότι έχουμε 15 κλουβιά, 15 πένες που παραπάνω θα κοστίζουν τώρα και όμω υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα διότι με τα παράνομα κλουβιά ε, κάποιοι θα μπορέσουν να έχουν ε, πλέον στην παραγωγή. Η Κομισιόν τι θα κάνει. Θα κάνει πίσω για να μπορέσει να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα. Δεν θα πρέπει να δοθούν περισσότερα περιθώρια. Επομένω, το ηθικό δίδαγμα είναι ότι αν η Ένωση ε, φτιάχνει μια οδηγία, τελικά πληρώνει ούτως ώστε να, να την αγνοούν οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε κύριε Ματράς. Και δίνει το στην κυρία Χέραντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το 2012 πρόκειται 400 παραγωγή να έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Περίπου 30% του έχουν παραγωγών στη χώρα και επομένω θα έχουμε 300.000 τόνου αυγά τα οποία δεν θα παράγονται πλέον. Και έχουμε επομένω σε αυτά τα 80 εκατομμύρια δύο, ε, και θέλουμε επομένω να καλυφθούμε με, πώς, με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εκεί όμως τα πρότυπα για την κολυμπλογή των ζώων είναι πολύ κατώτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω θα πρέπει να κινηθούμε με ευφύ τρόπο. Η οδηγία του 99 όσον αφορά τη, τα κλουβιά των ορνήθων ε, μας έδωσε κάποιες δυνατότητες και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή και να έχουμε επομένω ε, τέτοιες ευκαιρίες ε, και να ε, ανταγωνιστούμε αυτούς οι οποίοι έχουν κλουβιά πολύ πιο στενά, πολύ πιο μικρά. Πρέπει με αυτή την οδηγία να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες η παραγωγή. 600 εκατομμύρια ευρώ θα ανέβει το κόστος, αλλά μην ξεχνούμε τις συνέπειες οικονομικές για, το διατροφικό κλάδο γενικότερα. Παρακαλώ να ψηφίσετε ε, την τροπολογία μας, τη δεύτερη παράγραφο, την τροπολογία του ΕΛΚ. Εκεί ζητούμε να υπάρξει κάποια λύση για τις εκμεταλλεύσεις ε, των παραγωγών των υπευθύνων, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν ε, το, το, υλικό τους. Και θα έχουν σχεδόν ολοκληρώσει προσπάθειες το 2012. Να τους δώσουμε το περιθώριο τόσο ώστε να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους και έτσι να μην υπάρχει ε, αυτή η ανίκαιστος βλάβη για τις επιχειρήσεις και έτσι στην κοινοτική αγορά να αποφύγουμε την αύξηση της τιμής που θα βαρύνει τον καταναλωτή. Με αυτή την οδηγία να μπορέσουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στον κλάδο. Επίσης, να υπάρχει καλομεταχείριση των ζώων, αλλά και να μπορούν να έχουν λογικές τιμές καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. κυρία Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, <clears throat> θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα σαφώς ότι έχουμε αποφασίσει ήδη την κατάργηση της παλαιάς κοπής κλοβών. Είχαν η παραγωγή αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό και να διευθετήσουν τους κλοβούς τους και παραμένουν ακόμα 12 μήνες μέχρι <clears throat> το τέλος της προθεσμίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε όλες τις προσπάθειες ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με, τη νέα, με τις νέες προδιαγραφές κλοβών. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν επιτύχει να μεταγράψουν αυτή την οδηγία να βρεθούν ενώπιον ε, νομικών συνεπειών. παραδείγματο χάρη επιβολή προστήμων. Και εξάλλου, τα αυγά τα οποία έρχονται από κλωβούς που δεν είναι σύμμορφοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν θα πρέπει να μπαίνουν καθόλου στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρόντους. Η κυρία Ράιμερ, σε μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 12 χρόνια είναι γνωστό ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση η παλιή κλωβή για τις οτό και δεν θα είναι νόμιμη. Είναι πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν, χρειά, δεν τους έφτασαν 12 κράτη-μέλη για να μπορέσουν να προετοιμαστούν και να μεταγράψουν την οδηγία αυτή. Αυτό δείχνει πως από έλλειψη σωστής μεταγραφής και εφαρμογής μπορούν να προκύψουν προβλήματα. Ενώ τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα αντιμετωπίζουν σήμερα μια στρέβλωση ανταγωνισμού η οποία αντίκειται στι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Κομισιόν αντί να κάθεται στα αυγά τη να επιβάλλει κυρώσει στι χώρε οι οποίε δεν έχουν ε, εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό. Και από την 1η Ιανουαρίου 2012 τα αυγά αυτά τα παράνομα δεν πρέπει να μπαίνουν καν στην αγορά δεν πρέπει να, πληρώσουν την ύφη αυτοί που έχουν ε, μετατρέψει τους κλωβούς τους στις νέες προδιαγραφές να πληρώσουν το τίμημα της ολιγορίας ορισμένων κρατών μελών και ορισμένων παραγωγών. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τακτική η οποία θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Να μην εφαρμόζει κανείς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πάντα περιμένει κάποια παράταση. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται από όλους οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρχουν εξαίρεσεις για κανένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, όπως και όλες οι μητέρες, θέλουμε και την επιμερία των ζώων, αλλά και καλή ποιότητα αυγά. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων των αυγών. Ε, εγώ ξέρω απλώς ότι πρέπει να προστατεύουμε το κοτέτσι από τις, ε, ε, από τις αλεπούδες. Ε, και αυτό που θέλω είναι καλής ποιότητα αυγά. Ε, πρόκειται για μια ε, παραγωγή η οποία πλήρωσε πάρα πολύ ώστε να προσαρμοστεί στην ευημερία των ζώων εμείς σαν καταναλωτές της Βρετανίας έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και έχουμε πληρώσει ως παραγωγή πάρα πολλά χρήματα πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι οποίοι καλή την πίστη προσαρμόστηκαν στις ε, αρχές της οδηγίας. Thank you, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φόρτη, κυρία Μαγκίνες για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, ε, Επιτροπή για την ε, απάντησή της η οποία έστω και ατελής παρόλα αυτά μας δίνει πολλά θετικά στοιχεία. Εγώ βέβαια αμφισβητώ κυρίως τα αριθμητικά στοιχεία. Είπατε ότι 66% της παραγωγής είναι ελευθέρας βοσκής. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί οι πληροφορίες που έχω δεν είναι ίδιες. Νομίζω ότι λίγο Κάνετε επιλεκτική συλλογή των πληροφοριών ε, και των στοιχείων ε, και τα στοιχεία σας είναι, πώς να το πω, εμπλουτισμένα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα ήθελα να σας πω ότι θα, ίσως αν ήταν εύκολο να συμμορφωθεί κανείς με αυτήν την νομοθεσία και εάν πραγματικά και το υπογραμμίζω το πραγματικά ε, ε, ήθελαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ένα καλό σύστημα τότε θα πλήρωνα το αντίτιμο αλλά φαίνεται ότι πολλοί δεν θέλουν να πληρώσουν το αντίτιμο αυτό. Δεν έχω, ε, δεν έχω ούτε ένα αίτημα από καταναλωτή για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Και θυμηθείτε αγαπητοί μου συνάδελφοι έτσι έχουν τα πράγματα. Τούτων λεχθέντων είναι σημαντικό η νομοθεσία αυτή που έχει περάσει, που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο ε, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί. Πολλά χρήματα έχουν ε, ε, πέσει σε αυτήν την διαδικασία και ούτως ή άλλως πρόκειται για παραγωγή η οποία προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σας πω ότι στις αρχές του 2012 θα έχουμε 83 εκατομμύρια αυγά τα οποία, δεν, τα οποία θα είναι παράνομα. Δεν θα έχουν καν την απαραίτητη σφραγίδα. Και οπωσδήποτε για να καλυφθεί η απόσυρση των αυγών αυτών ε, θα πληρώσει τελικά το τίμημα ο καταναλωτής. Πάλι στο δικό του το κεφάλι θα πέσει αυτή η αναπόφευκτη κατάσταση γιατί αυτά τα αυγά θα βρίσκονται στην αγορά και επομένως χρειάζεται αποσαφήνιση. Όσον αφορά τώρα αυτούς που βρίσκονται στη μεταβατική φάση θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει οπισθοχώρηση. Μην ξεχνάτε το χρόνο σας λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά ξέρω ότι και ο Σάλεμος Άγνιου μίλησε πολύ περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιώδους σημασίας για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε περισσότερο χρόνο. Η κυρία Γκαρσία Πέρες για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Όπω βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να ε, τηρούνται οι διατάξει ακόμα και αυτέ που ακόμα δεν τέθηκαν σε ισχύ και αυτό έχει γίνει και σε άλλου κλάδου. Και έχουμε κάποιε προθεσμίε που πρέπει να, να τηρηθούν και γι' αυτό πάμε για ολομέλειε των 15 ημερών. Έχουμε τώρα ε, το, το, το, το, πόσο ε, αυξάνονται οι δαπάνες, το, το, κόστος, τα πάγια, οπότε θα πρέπει επομένως κάποιος να τηρήσει τα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί στην Ένωση. Επομένως όλα κατετείνουν στο ότι το 2012 την 1η Ιανουαρίου πάρα πολλοί παραγωγοί δεν θα έχουν μπορέσει 100% να, να τηρήσουν ό,τι χρειάζεται. Επομένως λέμε ότι θα λείπει ένα 30% της παραγωγής τόσο ώστε να καλυφθεί η αγορά και οι ανάγκες της. Επομένως το αποτέλεσμα είναι ότι τα φρέσκα αυγά θα είναι ε, πιο ε, ακριβά, θα πρέπει να αγοράσουμε απ' έξω αυγά και επομένως γι' αυτό ελπίζουμε ότι να υπάρχει αμοιβιότητα όσον αφορά αυτό το ζήτημα και τις σχέσεις με τρεις χώρες εν κατακλείδη ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιες παρεκκλήσεις για το 2012 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούσε να κάνει κάτι όσον αφορά να κάνει αυτό, το οποίο έκανε, αυτό που έκανε και με, με, με, με το πρόβιο και, και, και κρέας όσον αφορά την ε, σήμαση με ηλεκτρονικά μέσα και επίση να τηρηθούν ε, οι διατάξεις για την καλονταχείριση των ζώων. Πρόεδρος. Ο κύριο Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το ψήφισμα είναι σαφές το περιεχόμενο του. Καμία παρέκκληση, καμία εξαίρεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις για αυτούς που χρησιμοποιούν μη ε, αποδεκτές μεθόδους παραγωγής οών. Ορισμένοι είχαν 8 χρόνια για να προετοιμαστούν, άλλοι είχαν 5 χρόνια. Και αυτοί λοιπόν οι οποίοι είχαν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα προσαρμογής στη διάθεσή τους, βρεθήκαν σε μια θέση μειονεκτική. Πολλοί από αυτούς δεν κατανόησαν τι θα, συν, τι θα συμβεί όταν αγόραζαν φτηνούς κλοβούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση το, την παλαιά των 15 ετών. Στην πράξη όμως αυτό που θα γίνει είναι ότι θα υπάρξουν εισαγωγές αυγών από τρίτες χώρες που παράγονται σε απαράδεκτης μορφής κλωβούς. Δεν μπορούμε να πούμε σιγά τα ΟΑ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε μία λύση για αυτούς που δεν μπορούν να εξυγχρονίσουν τους κλωβούς τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 και γι' αυτό έχουμε καταθέσει και τις σχετικές τροπολογίες. Σύμφωνα με τους συντάκτες των τροπολογιών, η μεταβατική περίοδος ήταν γνωστή, ήταν καταγεγραμμένη μέσα στην οδηγία και η οριακή ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2012 δεν επιδέχεται τροποποίηση. Ελπίζω ότι αυτοί οι οποίοι θα υπερψηφίσουν το ψήφισμα αυτό θα υποστηρίξουν και την ιδέα ότι δεν πρέπει να δοθούν περαιτέρω μεταβατικές περίοδοι πέραν του 2013 σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές βάσει της κοινή αγροτικής πολιτικής <clears throat> γιατί ήδη οι τωρινές ε, διατάξεις ισχύουν μόνο μέχρι το 2013. Ευχαριστώ κύριε Καλινόφσκι. Ο κύριος Σταμπατζή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν κάνει τις απαραίτητες μετασκευές στους κλωβούς τους και αυτούς οι οποίοι παρέλειψαν να το κάνουν. Υπάρχει και μία ε, σύγκρουση μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ πολύ με τον κύριο Καλινόφσκι ότι τα παλαιά κράτη-μέλη είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για τη μετάβαση αυτή. Και κατάφεραν επίσης να πουλήσουν χρονιά τους παλαιούς κλωβούς του στα νέα κράτη-μέλη, γνωρίζοντα ότι και τα νέα θα έπρεπε να κάνουν αυτή την αλλαγή κλοβών. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τήρησαν απόλυτα τον, ε, την οδηγία αυτή και επομένως αυτή βρέθηκαν σε μια μειονεκτική θέση. Εμείς είμαστε <clears throat> πολλές φορές πολύ λιγότερο αυστηροί έναντι των εξαγωγέων από τρίτες χώρες από ότι είμαστε εναντίον των δικών μας γεωργών, τους οποίους με αυτόν τον τρόπο τους πλήττουμε. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες και δεν υπάρχουν καν και έλεγχοι. Και πάλι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει μια απόφαση η οποία δημιουργεί σε προβλήματα και μειονεκτήματα για μας. Ευχαριστώ Κύριο Παπαστάνκος για ένα, ένα μισή λεπτό. Κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της ε, Ένωσης υπέρ των παραγωγών οι οποίοι θα έχουν συμμορφωθεί με τις αυξημένε απαιτήσει που επιτάσσει η οδηγία. Παράλληλα όμως πρέπει να στηρίξουμε εκείνους τους παραγωγούς οι οποίοι δεσμεύονται με να συμμορφωθούν αδυνατούν όμως να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος προσαρμογής εντός της ταχθής σας προθεσμίας. Προβλέπετε ότι τα μη συμφώνως προς την ομοθεσία παραχθέντα προϊόνα, προϊόντα δεν θα μπορούν από 1η Πρώτου 2012 να διατίθενται νομίμως και να αποτελούν αντικείμενο ενδοκινοτικού εμπορίου. Παράλληλα όμως θα εξακολουθήσουν να εισάγονται από τρίτες χώρες προϊόντα ελαστικότερων προδιαγραφών προστασίας των ζώων. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κινδυνεύουν να τεθούν εκτός παραγωγής πολλές μονάδες της Ένωσης, χάρη της αυξημένης προστασίας των ζώων, θα εισάγονται προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία δεν θα πληρούν ούτε καν τις προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα στην Ένωση. Ναι, να προστατεύσουμε την ευζοία, το animal welfare, να προστατεύσουμε όμως και τον ευρωπαϊκό κοινωνικοπαραγωγικό ιστό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Mr. is next. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Επίτροπε, αν και όλοι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θα πρέπει να σέβονται την κοινωνική νομοθεσία και να προβαίνουν έγκαιρα στις αναγκαίες προσαρμογές, εκτιμάται ότι το 30% των αυγοπαραγωγών δεν θα έχει προβεί σε αυτές μέχρι τη 1 Πρώτου του 2012. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα που μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει να πείσει τους παραγωγούς ότι αυτό σημαίνει όφελος για εκείνους και μια πολιτική που δεν έχει πείσει τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους να την περιφρουρήσουν είναι δύσκολο να επιτύχει όποια και να είναι τα μέτρα αστυνόμευσης που θα επιβληθούν πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συνέδεε το κόστος της επένδυσης με το όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή από τη χρήση των εμπλουτισμένων κλοβών θα έπειθε περισσότερο του παραγωγούς για την υιοθέτηση του μέτρου. και βέβαια μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί παρά να κατοχυρώνει τη διακριτή διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού προϊόντος με βάση χαρακτηριστικά ποιότητας ασφάλειας και ευζοίας των ζώων προκειμένου να το προστατεύσει εναντί αθέμητου ανταγωνισμού με άνισους όρους από τρίτες χώρες έτσι όπως φοβούμαστε ότι πρόκειται να συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαβία παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της ευζοίας των ζώων είναι ένα θέμα το οποίο εδώ στην Ολομέλεια επανειλημμένα έχουμε αντιμετωπίσει και πιστεύω ότι έχει επιλέξει το Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο έχει κάνει, λοιπόν, έχουν κάνει τα τρία όργανα μια σταθμισμένη και ισορροπημένη επιλογή. Δεν μπορούμε τώρα να επιστοδρομήσουμε. Οφείλουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Ε, στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη και αναλογιζόμενοι και τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους αυτούς ε, τους γεωργούς ε, που έχουν προσαρμόσει ήδη την διαδικασία παραγωγής τους. Είναι σαφές ε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω περίοδος χάριτος έτσι ώστε να υπάρξει μετάβαση προς ένα υπεύθυνο σύστημα όσον αφορά την ευζοία των ζώων. Έχουμε την ευθύνη να σκεφτούμε όλους αυτούς που έχουν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία μετάβασης και μάλιστα το πράττουν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, περίοδο κρίσης η οποία δυσκολεύει κάθε επένδυση θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ακριβώς στο ζήτημα της μετάβασης, δηλαδή το ζήτημα όλων αυτών των κτηνοτρόφων που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους την ευζοία των ζώων, αλλά δεν, το, δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μετάβασης. Και πιστεύω ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο της κρίσης θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή προς τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Βλέπω ήδη ότι σηκώνονται αρκετά χέρια. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Νικολέσκου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γενικεύουμε και να γενικολογούμε. Αλλά, ε, ξέρετε, στη Ρουμανία και η Βουλγαρία μπήκαν στην Ένωση πριν από τρία χρόνια μόλις και βεβαίως θα πρέπει και να τηρούνται οι νόμοι. Παρακαλώ να επιψηφίσετε την ε, τροπολογία για την παραγραφό 2 του ΕΛΚ. Έχουμε πάρα πολλού ε, παραγωγούς που προσπαθούν να συμμορφωθούν, γίνονται επενδύσει, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά ε, πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρωθούν, αλλά και γι' αυτό δεν πρέπει όμω να του τιμωρήσουμε πάρα πολλοί έχουν αρχίσει να βελτιώνουν την, ε, το υλικό τους και προσπαθούν να τηρήσουν επομένω τις συνθήκες που έχουν προβλεφθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ο κύριος Μπρόνς έχει το λόγο. Οι παραγωγές στο Ενωμένο Βασίλειο έχουν επενδύσει και πολλά χρήματα και έτσι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί λόγω αυτής της οδηγίας. Ξέρετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρήσει τον νόμο, όμω θα έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό για κάποιε χώρε οι οποίε δεν θα το κάνουν το ίδιο ή θα πάρουν κάποιο είδου εξαίρεση όσον αφορά την ε, υλοποίηση. Και επομένω θα ισχύσουν διαφορετικά πράγματα σε, σε κάθε χώρα στην Ευρώπη των 27. Θα έπρεπε επομένω να υπάρχει κάποιο είδου αποτροπή. Όταν υπάρχει τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να ε, την εφαρμόζουν όλοι και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Θα έπρεπε να μην επιτρέπεται να εξάγουν αυγά οι χώρες που δεν θα τηρήσουν την ε, οδηγία. Και οι παραγωγοί ζητούν την προστασία κατά του αθέμητου ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Μπορείς, ευχαριστώ και τώρα κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα θα ήθελα να επαναλάβω ότι θεωρώ ότι οι οδηγίες υπάρχουν για να εφαρμόζονται και αυτό ισχύει και για την οδηγία του 1999. Και επίσης η απασχόληση της, η της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευζοία των ζώων είναι μια από τις βασικές σημαίες και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται <clears throat> για μια οδηγία η οποία οδήγησε σε πολύ μεγάλο κόστος. 30% παραπάνω για κάθε κότα στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη. Όταν έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μικρά κεφάλαια, έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες εμπόδισαν τον εξυγχρονισμό πολλών επιχειρήσεων και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν και μόνο αυτές που ξεκίνησαν την προσαρμογή να φέρουν σε πέρα σε αυτή την προσαρμογή. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλβέστρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Επίτροπε, κανένας από εμά δεν θέλει να αμφισβητήσει την ανάγκη ε, σε μια οδηγία ε, η οποία ήδη είναι παλαιά ούτε να αμφισβητήσει τη σοβαρότητα του θέματος. Το κυριότερο ζήτημα βεβαίως ήταν ε, η ευζοία των ζώων, αλλά βεβαίως η οδηγία και η εφαρμογή της θα πρέπει να βασίζεται και στην λογική. Πρώτα απ' όλα, από το 99 μέχρι τώρα ε, ε, μεσολάβησε μια πολύ βαθιά οικονομική κρίση η οποία ε, δημιούργησε, προκάλεσε μάλλον πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και γι' αυτό οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. 1η Ιανουαρίου 2012 λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούν, αλλά αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να βγουν από την αγορά και από την παραγωγική διαδικασία. Βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους ε, ε, παραγωγούς αλλά έτσι τους σπρώχνουμε έξω από την Ευρώπη. Μία στιγμή, σε μία περίοδο μεγάλης κρίσης όπου μεγαλώνει η ανεργία, όπου αυξάνονται τα ελλείμματα, όπου δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά για επιπλέον επενδύσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να οδηγήσουν την Επιτροπή στο να ξανασκεφτεί λίγο το θέμα της παράτασης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλβέστρη. Η κυρία Ντότσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως τόνισαν πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, η προστασία των παραγωγών που έχουν δαπανίσει πολλά χρήματα για να αλλάξουν τους κλωβούς τους είναι κάτι απαράγραπτο και είναι καθήκον της Κομισιόν σε αυτό το στάδιο. Αλλά πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αναγνωρίσει και το έχω τονίσει και σε πολλούς από τους γεωργούς που ε, με τους οποίους μίλησα που δεν έχουν τα χρήματα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία να επενδύσουν για τη μετασκευή αυτών των κλοβών να υπάρξει κάποια ε, ρύθμιση και για αυτούς. Το θέμα της ετικετοποίησης ή της φράγησης των αυγών είναι σαφές για μένα ότι δεν πρόκειται να έχουμε κανένα όφελος με περαιτέρω επίθεση σφραγίδων. Δεν πρόκειται να κάνουν οι καταναλωτέ κάποια διάκριση μεταξύ αυτών των αυγών και των εισαγωμένων παραγωγών χάρη των αυγών Τουρκία. Για του λόγου όλου αυτού θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να μα πει αν θα μπορούσε να εξασφαλίσει να υπάρξει μια εξαίρεση. Οι εταιρείε στη δική μου περιοχή που εισάγουν αυγά από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υποχρεωμένες να μην παίρνουν αυγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παίρνουν αυγά τα οποία θα έχουν παραχθεί κάτω από λιγότερο αυστηρούς ελέγχους. Ευχαριστώ κύριε Αντώτ. Κύριο Σκερεύσκη. Σας ευχαριστώ. Είναι σαφές από τη συζήτηση ότι η ε, οι γεωργοί και οι εκτινοτρόφοι θα πρέπει να σεβαστούν την οδηγία του 1999. Καταλαβαίνουμε τη θέση αυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει στον εξυγχρονισμό των κλοβών. Δεν είναι ο στόχος να δώσουμε σε ορισμένου μονάχα χρόνο <clears throat> προσαρμογής. Αυτό το πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε σε όλους τους γεωργού τον ίδιο χρόνο που θα τους επιτρέψει να εξασφαλίσουν τα κριτήρια και τι προδιαγραφέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή, η παράνομη παραγωγή αυγών φαίνεται μια ενδιαφέρουσα προοπτική αλλά θα πρέπει εμείς να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην προστασία των καταναλωτών. Γιατί όμως να υπάρχει σεβασμός των καταναλωτών σε ορισμένε περιοχές και όχι σε άλλες. Εγώ υποστηρίζω οποιοδήποτε μέτρο το οποίο θα δώσει βοήθεια σε όλους τους γεωργούς στα κράτη-μέλη, γιατί ξέρω ότι οι Γεωργοί βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη εισοδηματική κατάσταση αυτή τη στιγμή και κρίμα που δεν συμφωνούν όλοι μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές για όλους μας πιστεύω ότι η ευζοία των ζώων και η υγεία των ζώων με την οποία συνθέεται η ανθρώπινη υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στην ΣΤΟΑ, στην ε, ε, Επιτροπή που εξετάζει επιστημονικές και τεχνολογικές επιδεολογίες εξήτασε ορισμένες δυνατότητες με τις οποίες μπορεί να βελτιωθεί η εκτροφή των οτόκων ονήθων. Θα ήθελα ε, γι' αυτό να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο, ιδίω στα πλαίσια του 8ου προγράμματος πλαίσιου για τα τρόφιμα να ενισχυθεί ο τομέας αυτός ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ασφάλεια των τροφίμων και την ευζοία και υγεία των ζώων και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες της Ευρώπης την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρούμπ. Κύριε Μακίνες και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να θίξω και άλλα δύο σημεία και δεν πρόλαβα προηγουμένως. Το θέμα των ε, αυγών είναι σαφές, αλλά υπάρχει και μία ε, διαδικασία παραγωγής για τα αυγά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ε, στην υπόλοιπη διατροφική αλυσίδα για άλλες παραγωγές κτλ. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί όλο και περισσότερος είναι ο αριθμός των αυγών που τελικά καταλήγουν στην μεταποίηση Επίσης υπάρχουν προϊόντα τα οποία βασίζονται στο υγρό αυγό ή στο αυγό σε σκόνη και ε, πιστεύουμε ότι και εκεί θα πρέπει να δούμε από πολύ κοντά τα πράγματα. Ε, φοβούμαστε ότι θα υπάρχει ένα παράλληλο, ένα παράλληλο σύστημα παραγωγής ε, και επομένως φοβούμαστε ότι όταν θα ξεκινήσει το νέο σύστημα κλοβών παρόλα αυτά θα παραμείνει στην αγορά και θα παράγει αυγά ένα παράλληλο σύστημα κλοβών και αυτό μας απασχολεί πολύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λυθεί σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκίνες. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει στο Catch the Eye. If that's not the case, I give the floor. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βασιλείου η οποία θα κλείσει τη συζήτηση και θα απαντήσει ενδεχομένω κάποιε ερωτήσει που έχετε υποβάλει. Πρόεδρε, ευχαριστώ λέει κυρία Βασιλείου. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε συνένεση για το θέμα μας. Άκουσα κάποιοι βουλευτές να ζητούν να μην υπάρξουν παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις. Όμως από την άλλη μεριά, από άλλους, άκουσα το αντίθετο, να θέλουν χορήγηση παρεκκλήσεων. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από ποια χώρα προέρχεται ο καθένας και σε ποια φάση βρίσκεται κάθε χώρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Να σας πω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω, από 1η Πρώτου 2012 οι συμβατικοί κλοβοί θα πρέπει να αντικατασταθούν με το νέο τύπο κλοβών ή εναλλακτικά συστήματα. Οπότε, τα αυγά από του συμβατικού κλοβού δεν πρόκειται να επιτρέπεται να τίθενται σε εμπορία μετά την 1η του 2012. Αυτή είναι η θέση μας. Καταβάλουμε δε πάσα δυνατή προσπάθεια να βοηθήσουμε τις χώρες να συμμορφωθούν με την οδηγία. Και τι κάνουμε συγκεκριμένα. Πρώτα πρώτα, ενθαρρύνουμε την ε, θέσπιση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων με την εμπλοκή των ενδιαφερομένων. Και βεβαίως να προβλέπονται και κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με την οδηγία. Δεύτερον, βοηθούμε την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε ανταλλαγή των ε, αρίστων πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και έχουμε και κάποιους εμπειρογνώμονες που βοηθούν στην υλοποίηση της οδηγίας. Επίσης, οργανώνουμε συναντήσεις με εμπλεκόμενους, όπως σας προανέφερα, στις 19 Ιανουαρίου του 2011 θα έχουμε μια τέτοια μεγάλη συνάντηση. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των κρατών μελών και εκεί πρόκειται να συζητήσουμε το πώς έχουν τα πράγματα. Και να δούμε πώς μπορούμε τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε κάποια κρατημέλη που ακόμα δεν έχουν τους αθιές τους να τις ολοκληρώσουν ε, μέχρι το τέλος του επομένου έτους. Αυτή είναι η θέση μας. Και ενή περιπτώσει μετά την πρώτη η Πρώτη 2012 ακόμα υπάρχουν αυγά τα οποία δεν θα παράγονται συμφώνως τον νόμο δεν θα μπορούν να τίθενται σε εμπορίο και σε κάθε περίπτωση που θα έχει αποδειχθεί παραβίαση της οδηγίας θα ληφθούν τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία δηλαδή θα αρχίσει η διαδικασία επί παραβιάση του κοινωτικού δικαίου ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της κοινωτική νομοθεσίας. Επίσης, ε, σαν εναλλακτική λύση, προσπαθούμε να δούμε πώς θα φρενάρουμε την παράνομη θέση σε εμπορία αυγών που δεν έχουν παραχθεί συνόμως μετά την προηγούμενη άκουσα και κάποιες παρατηρήσεις από ε, κάποιους αγορητές και όλα όσα είπατε θα τα διαβιβάσω στον Επίτροπο Ντάλη ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα τα λάβει υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Λέει ο Πρόεδρος. Κυρίες συνάδελφοι, έχουν ζητηθεί ε, να συζητήσουμε και άλλα τέσσερα θέματα. Επομένω, εδώ πέρα τελειώνει αυτή η συζήτηση. Θα κάνουμε όμω ε, την ψηφορία και μετά συνεχίσουμε. 12 η ώρα αρχίζει η ψηφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι ανορθόδοξο το να ζητεί κάποιο το λόγο όταν κλείσει τη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σα πω ότι ε, μα χρεοποιούν τα, τα όσα είπε Επίτροπο. Όμω ε, αυτό το, το, το συμπέρασμα ότι εμεί είμαστε διχασμένοι για το θέμα μα δεν είναι δικαιολογημένο. Οπότε παρακαλώ με κάθε σεβασμό να κάτσει η κυρία Επίτροπο και να δει τη, τα αποτελέσματα τη τελική ψηφοφορία πριν διαμορφώσει άποψη για το κατά πόσο είμαστε διχασμένοι. Και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βεβαία ότι η κυρία Επίτροπο θα το κάνει αυτό. Ε, σταματούμε λοιπόν μέχρι τις 12, οπότε θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. 12 το μεσημέρι. Λοιπόν. Point of order. Sorry, I didn't see you. Thank you, President. Can I first of all support... Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω, θα στηρίξω την Έστερ σε αυτά που είπε προηγουμένως. Επίσης, πραγματικά δεν πίστεψα ούτε μία στιγμή ότι το, το, σώμα είναι μοιρασμένο. Και επίσης ε, ε, όταν λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία επιπλέον σήμανση, ε, τι εννοεί ακριβώς γιατί υπάρχουν τα αυγά αυτά τα οποία θα παραχθούν ε, παράνομα και τα οποία δεν θα μπορούν να φέρουν αυτή τη σήμανση. Πρόεδρος, δυστυχώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Ε, έπρεπε να είχατε μιλήσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κύριε Ρούμπιχ, διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, διοργάνωση των εργασιών μας που εξασφαλίζει ότι υπάρχει και κάποιο διάστημα στην Ολομέλεια ένα τέταρτο διάλειμμα μέχρι την αρχή των ε, ψηφοφοριών και αυτό εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει χαοτική κατάσταση στην Ολομέλεια. Έτσι πρέπει να είναι πάντα, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ.